έχει προβεί στην ε, επαλήθευση της εντολή, ε, γύρω Ντιτιέ και Τζοάνα και ε, πρότεινε να επικυρωθεί η εντολή τους από 1η 12 17 και 30 Ιανουαρίου 2018 αντιστοίχως.